θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα σε ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την ανοικοδόμηση και τον εκδημοκρατισμό του Μαλή. δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές, πρώτα στην κυρία Ζολή για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, η ανοικοδόμηση του Μαλή και ο εκδημοκρατισμός είναι τεράστια θέματα. Θα συγκεντρώσω όμως σε τρία θέματα την προσοχή μου κυρίως στο ρόλο μας στη διαδικασία ανοικοδόμησης, στην ειδική φροντίδα για τα θύματα βιασμού, όπως επίσης και στην οικονομική βοήθεια. Δεν νομίζω ότι με την παρέμβαση που έγινε λύθηκε ε, το πρόβλημα του Μαλή. Προφανώς απαιτείται να υπάρξει μια ε, νόμιμη εξουσία στην χώρα αυτή για να ανοικοδομηθεί αλλά ακόμα όλα αυτά δεν είναι πολύ ε, αποτελεσματικά και είναι πάντα εύθραυστα και δεν μπορεί να γίνει εκλογική διαδικασία ή ειρηνική. Πάρα πολλές γυναίκες κατά τη διάρκεια του φρικτού πολέμου βιάστηκαν ή ε, αναγκάστηκαν να παντρευτούν με βία, εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, οικογένειες που πρέπει να τις ακούσουμε και να τις βοηθήσουμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις συνδράμει μέσω των μη κυβερνητικών οι οποίες όμως δεν, οργανώσεων που δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα. Στη βία αντίθεται και το θέμα της ημερομηνία των εκλογών όπως επίσης και της ψήφου των προσφύγων και έχει ε, επιλεγεί λανθασμένη ημερομηνία στην αρχή του Ραμαζανιού και στην εποχή των βροχών. Λοιπόν, ας μην πολλαπλασιάζουμε τα εμπόδια τα οποία έτσι και αλλιώ υπάρχουν. Το θέμα είναι να διασφαλίσουμε την παροχή των βασικών υπηρεσιών και την ανοικοδόμηση της, των υποδομών της χώρας. Αυτό θα βοηθήσει τον λαό να δει την προσπάθεια που γίνεται με διαφορετικό μάτι. Η γαλλική παρέμβαση μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε στο διάλογο και να ακούσουμε όλες τις συνιστώσεις της ε, κοινωνίας του Μαλή, ακόμα και αυτές που ασκούν σκληρή κριτική. Το μέλλον του Μαλή ανήκει στους κατοίκους της. Δεν θα επιλέξουμε εμείς ε, τους ε, συνομιλητές μας. Η παρέμβασή μας, η οποία κρίνεται σαν απελευθερωτική από πολλούς κατοίκους, θα παρεξηγηθεί για νέα πικιοκρατία. Θα πρέπει να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντανζάν, τρία λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι μιλώ και εκ μέρους του Έλμερ Μπρόκ, που είναι ε, και εκείνο συντάκτη αυτού του ψηφίσματος, αλλά δεν, μπορεί να είναι, δεν μπορούσε να είναι ε, απόψε μαζί μας. Ναι, καταρχήν διαπιστώνουμε ότι αυτή η συζήτηση φτάνει σε μια στιγμή σημαντική για το Μάλι. Είναι μια συζήτηση που δυστυχώς θα ήταν πολύ χρήσιμο να την είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα. Και όταν λέω νωρίτερα εννοώ χρόνια νωρίτερα. Γιατί δεν πρέπει να παραλείψουμε να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη-μέλη και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011, πάνε πάνω από δύο χρόνια, είχαν αποφασίσει για μια στρατηγική ανάπτυξη για το Σαχέλ. Αν είχε εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική, σίγουρα δεν θα βρισκόμασταν σήμερα στο σημείο που βρισκόμασταν να πρέπει να, έχουμε, να προτείνουμε ένα ψήφισμα το οποίο μιλά για τέτοιες πολιτικές ασφάλειες και στρατηγική σε ένα πλαίσιο πολύ πιο δύσκολο από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Σήμερα πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο κατεπηγόντως και όταν ε, κάνουμε κάτι με επίγοντα χαρακτήρα ποτέ δεν ε, είναι προς όφελός μας. Η κυρία Ζολή πολύ σωστά μίλησε για την εκλογική διαδικασία. Βεβαίως χρειάζονται εκλογές, βεβαίως ε, το καλύτερο πράγμα είναι οι εκλογές για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί το τοπικό καθεστώς και οι φορείς με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε επί τόπου και που τελικά είναι αυτοί που θα είναι υπεύθυνοι για το, για το μέλλον της χώρας τους. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε γιατί αν ένα εκλογικό εκλογικό ε, σύστημα, αν ε, μια εκλογική διαδικασία ε, γίνει με τρόπο ασφαλμένο για τεχνικούς λόγους, αν οι εκλογές δεν διεξαχθούν σωστά, μπορεί να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την νομιμοποίηση των διαφόρων παραγόντων. Και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε για τη βιασύνη με την οποία πιέζεται αυτή η εκλογική διαδικασία. Υπάρχουν δύσκολες συνθήκες και όσον αφορά την ασφάλεια. Και εδώ χαιρετίζω το έργο του Γαλλικού στρατού μαζί με τους Αφρικανούς συμμάχους και πρέπει επίσης ε, να χαιρετήσουμε και το έργο της ε, Ευρωπαϊκής Αποστολής, της EUTM ε, που ασχολήθηκε με την εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει και τη συνέχεια και τη διάρκεια γιατί ο στρατός στο Μαλή χρειάζεται κάτι παραπάνω από εκπαίδευση και κατάρτιση. Χρειάζεται μια νέα δημιουργία, μια αναδιάρθρωση. Χρειάζεται ένα στρατός που να είναι πιστός προς τις αρχές, ένας στρατός που να ακολουθεί την πολιτική των θεσμών της χώρας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο εδώ. Και θα πρέπει επίσης ε, και εδώ και στις Βρυξέλλες να δούμε τα διδάγματα από τα προβλήματα που υπήρξαν και από τις ελλείψεις που υπήρξαν στη φάση πριν από την σύραξη. Και θα πρέπει ε, όλοι να ασχοληθούν για να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική στο Μάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Πίμπαξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω μαζί σας για το Μαλί. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό το θέμα εν ώψη των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν μετά από ένα μήνα περίπου. Επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη πρόκειται να αναλάβουν τη διεθνή αποστολή στο Μαλί που μέχρι τώρα ε, βρισκόταν υπό αφρικανική ηγεσία. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσεις που τέθηκαν, θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη έχει ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κρίσης ε, που απείλησαν σοβαρά και το Μαλί και τη γενικότερη περιοχή του Σαχέλ. Και μάλιστα δράσαμε σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ του 2011. βέβαια ε, η πολιτική αυτή υπόψη τα δικαιώματα των ε, νόμιμων αρχών και μάλιστα με συντονισμένο τρόπο μέσω της συμμετοχή μας ε, στην ε, ομάδα, στη Διεθνή Ομάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης και με τις διμερείς προσπάθειες των κρατών μελών δώσαμε το παρόν στο Μαλί. Και μάλιστα και πριν το πραξικόπημα της 22ης Μαΐου του 2012. Επιπλέον προσφέραμε σημαντική έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 112 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ αλλά και με διμερή βοήθεια. Η Ευρώπη έχει, αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο τμήμα της διεθνούς προσπάθειας για την υποστήριξη στο Μαλί. Πέραν της, Ευρω... της επιχείρησης Ερβάλ, της, ε, της ε, ε, διευκόλυνσης για την Αφρικανική ειρήνη και την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Αφρικανικών δυνάμεων, κοβάς, δώσαμε 50 εκατομμύρια. Επίσης έχουμε την αποστολή EUTM για την κατάρτιση και εξάσκηση του στρατού του Μαλή. Και μάλιστα ζητήσαμε εκπόνηση οδικού χάρτη για το Μαλή που επιτέλους υιοθετήθηκε στις 29 Ιανουαρίου και μάλιστα προσφέραμε και υποστήριξη για την εφαρμογή του. Είμαστε ο βασικός εταίρος του Μαλή εδώ και δεκαετίες και μάλιστα ο κύριος διεθνής διαφερόμενος και συμμέτοχος στην ανακοδόμηση της χώρας. Ο σημαντικός μας ρόλος φάνηκε στις 15 Μαΐου του 2013 στην Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου των Δωρητών με συμπροεδρία Μαλή, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γαλλίας έχουν δοθεί υποσχέσει για πολύ σημαντικά οικονομικά μέσα ύψους 3,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρώπη μάλιστα προσφέρει 1,4 δισεκατομμύρια, από τα οποία 848 εκατομμύρια προέρχονται από τα κράτη-μέλη και 523 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές δεν είναι μόνο συμβολικές υποσχέσεις, αλλά ανταποκρίνονται στο σχέδιο δράσης που έχει ετοιμάσει το Μαλί. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εφαρμόζει μια συνολική προσέγγιση και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Ε, ανθρωπιστική βοήθεια, μέσω για τη σταθερότητα, θεματικά περιφερειακά προγράμματα και φυσικά προσπάθειες για τη δημιουργία υποδομών. Θέλουμε να συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση της χώρας, την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τον κατευνασμό της κρίσης που μαστίζει το Μαλί από το 2012 και μάλιστα ξεκινήσαμε κάποια προγράμματα ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση και θα έχουμε και επιπλέον παρεμβάσεις φέτος με βάση το σχέδιο ανάκαμψης του Μαλή για το 2013-2014. Μάλιστα η ύπατη εκπρόσωπο, όρισε και ειδικό εντεταλμένο της ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαλί που θα παίξει ε, σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των συνομιλιών στο Μαλί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών προκειμένου να ανακτηθεί ο έλεγχος του κράτους ε, και του συνόλου της επικράτειας, ιδιαίτερα της περιοχή Κιντάλ στο βορρά. Ε, είμαστε παρόντες σε όλες τους τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στον οδικό χάρτη του ΟΜΑΛ. Υποστηρίζουμε την μεταρρύθμιση του στρατού υπό δημοκρατικό έλεγχο, υποστηρίζουμε την Διεθνή Επιτροπή Επανασυμφιλίωσης και στηρίζουμε τις εκλογές με μία αποστολή παρατήρηση εκλογών με επικεφαλή στο Λουί Μισελ. Η διπλωματική μας παρουσία και η συνολική μας αξιοπιστία στην περιοχή αυτή είναι πολύ καλές και παρά τις επικρίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσαρμόστηκε με πολύ άμεσο τρόπο σε μια ραγδαία εξελισσόμενη κατάσταση. Και μάλιστα το μέσο και του πακέτου σταθερότητας των 20 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε κάποιες έκτακτες ανάγκες και ε, να συμβάλλουμε στη διαμεσολάβηση. Η βοήθεια μάλιστα στη Μαυριτανία και τον Ήγηρα έχουν προσαυξηθεί κατά 25 εκατομμύρια το Μάιο. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η ε, μη στρατική αποστολή UCAP της ΚΕΠΑ έχει ξεκινήσει τη δημιουργία υποδομών στον Ήγηρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε και την ε, την Επιτροπή του Σαχέλ για την Ασφάλεια με πρωτοβουλία Νίγηρα, Μαυριτανία και Μαλή. Παρ' όλα αυτά το πιο δύσκολο τμήμα είναι μπροστά μα ακόμα και στο Μαλή και στην ευρύτερη περιοχή και χρήζει τη αδιάσπαστη προσπάθεια και προσοχή μα. Στο Μαλή η ανοικοδόμηση είναι μια πολυσχηδή πρόκληση και σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση των τοπικών φορέων και παραγόντων να πραγματοποιήσουν πρόοδο σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει τη διακυβέρνηση. Βέβαια θα πρέπει να παράσχουμε με αποτελεσματικό τρόπο την διεθνή βοήθεια γιατί τις τελευταίες δύο δεκαετίες έγιναν πολλά λάθη και οι προσφορές των δωρητών δεν είχαν τον αναμενόμενο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη και μάλιστα η μεταρρύθμιση του δομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και η εμβέδωση του κράτους δικαίου έχουν ευρελική σημασία και μάλιστα οι ρυθμίσεις για καταμερισμό του βάρους διεθνώς δεν έχουν προσδιοριστεί αλλά η Ευρώπη με τα κράτη-μέλη θα αποτελέσει σημαντικό παίκτη στην προσπάθεια δημιουργίας υποδομών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Σταθερότητας, καθώς και με τη δράση της ΚΕΠΑ. Η παρασυμφιλίωση στο Μάλι επίση θα είναι περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Έχουμε κινητοποιήσει μέσα για να βοηθήσουμε την Εθνική ε, Επιτροπή Διαλόγου και μάλιστα ε, έχουμε και ένα ε, πρόγραμμα για την προώθηση της ειρήνης. Μια επιτυχή σε παρασυμφιλίωση όμως προϋποθέτει δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών να βρουν μια λύση. Και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών που γίνονται στο Μαλί με τη διευκόλυνση του δικού μας ειδικού εντεταλμένου και της αντιπροσωπείας του. Να αναφερθώ και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι οι αρχές του Μαλή ευαισθητοποιούν το στρατό για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αξιοπρόσεκτο. Αλλά θα πρέπει να επαγρυπνούμε για να αποφύγουμε τα έκτροπα από όλε τι πλευρέ. Ε, χρηματοδοτούμε και αποστολές, ε, αφρικανικές αποστολές παρατηρητών. Αλλά πολλές φορές γίνονται παραβιάσεις που διακυβεύουν την επανασυμφιλίωση. Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουμε προστασία που χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά το περιφερειακό επίπεδο, διασυνοριακή συνεργασία για την ασφάλεια αποτελεί σημαντική πρόκληση, όπω ε, ε, φάνηκε από τι πρόσφατε επιθέσει στον Ήγηρα και την Αργερία. Πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμη όμω ε, στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τη διαφθορά. Δεδομένη κατάσταση στη Λιβύη, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί ένα περιφερειακό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση της Σαχάρα στην περιοχή του Σαχέλ, κάτι που λείπει τώρα. Θέλουμε ένα φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ βορειοαφρικανικών χωρών και χωρών Σαχέλ μαζί με διεθνείς εταίρους, κάτι που είναι σημαντικό για άμεσα θέματα ασφάλειας αλλά και πιο μακροπρόθεσμες κοινωνικο-οικονομικές ε, προκλήσεις. Πιστεύω ότι συμβολή μα και η συνδρομή μας στο Μαλί είναι πολυσχηδή και ευρύτατη. Δεν μπορούμε όμως να υποκαταστήσουμε την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει από το ίδιο το Μαλί που θα πρέπει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Οι εξελίξη των τελευταίων μηνών μας ε, έδωσαν τι διαβεβαιώσει ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και το ίδιο το Μαλί για να ξεπεραστεί η κρίση και να διορθωθούν τα σφάλματα που έγιναν. Θα πρέπει όμως το ίδιο το μαλλί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Εμείς ε, χορηγούμε την απαραίτητη βοήθεια και συνδρομή όπου χρειάζεται και μάλιστα η συνδρομή μας είναι αξιοπρόσεκτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματων των ομάδων. Ο Πρέντα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την επικαιρότητα στην Ουάγκα υπό την προεδρία του Καμπαορέ, του Προέδρου Καμπαορέ, ωραίος. Υπεγράφει, μη υπογράφεται μια συμφωνία για την κατάσταση στο Κιντάμ. Και υπογραμμίζουμε τι σημασία έχει η υπογραφή για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, γιατί αλλιώς οι εκλογές θα τεθούν σε κίνδυνο και η κατάσταση παραμένει εύθραστη. Πάντως σας μείνουμε αισιόδοξοι και σε επανέλθουμε στο κεντρικό θέμα της συζήτησής μας, το θέμα της ανοικοδόμησης, γιατί όπως ακούστηκε υπήρξε μια στρατιωτική παρέμβαση, επιτυχεστάτη, επενέσαμε τη γαλλική προσπάθεια επανειλημμένα και απ' την άλλη υπάρχουν και υποσχέσεις για βοήθεια. Η διάσκεψη μαζί για το Μαλί, για το νέο Μαλί, οι ανάγκες της χώρας είναι τεράστιες. Οι πόροι της κυβέρνησης του Μαλή μειώθηκαν κατά 30% μετά το πραξικόπημα του 12. 1,5 εκατομμύριο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Λείπουν οι ιατρικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση στο βορρά, και ένα εκατομμύριο κάτοικοι της χώρας υποφέρουν από την πείνα. Η πρόκληση είναι μεγάλη λοιπόν και η Ευρώπη κάτι θα πρέπει να κάνει στη συγκεκριμένη βέβαια συγκύρια. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες 1,5 λεπτό η κυρία Γκόμες. Ο εκδημοκρατισμός του Μαλή εξαρτάται από το, την κατάπαυση της βίας και του πυρός και φυσικά από, τις, από την επιθυμία επανασυμφιλίωσης. Διερωτώ με όμως, μια τέτοια σπευσμένη εκλογική διαδικασία και χωρίς να ασφάλεια, αν θα έχει θετικό αντίκτυπο στη μετάβαση. Γιατί η σταθεροποίηση της χώρας προϋποθέτει τεράστιες προσπάθειες επανασυμφιλίωσης εθνικής, πολιτικής και κοινωνικής, ε, με συμμετοχή του έθνους του ΑΡΕΓ, με συμμετοχή όλων των στρωμάτων της κοινωνίας του Μαλή. Και ο αποφασιστικός ρόλος που δίνονται και οφείλουν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στη διαδικασία αυτή, προϋποθέτει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους και να δοθεί προβολή στο ρόλο τους, γιατί οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Επίση, θα πρέπει να εξαρθρωθούν τα εγκληματικά κυκλώματα και τα τρομακρατικά, γιατί αποσταθεροποιούν όχι μόνο το Μαλί, αλλά όλη την περιοχή του Σαχέλ. Και για να παραμείνει το Μαλί στο δρόμο του εκδημοκρατισμού, θα πρέπει οι αρχέ του Μαλί, με την ε, στήριξη τη ε, διεθνού κοινότητα και ιδιαίτερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να δεσμευτεί για την κοινωνική ανάπτυξη τη χώρα. Γιατί αν δεν ικανοποιηθούν οι θεμελιώδει ανάγκε του λαού, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή η ρυθμή ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλή, δεν θα μπορέσει το Μαλί να εξασφαλίσει μια κατάσταση και ένα πρόσφορο έδαφος για να εξυγχρονιστεί ε, πολιτικά και οικονομικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να επενδύσει σε μια στρατηγική ολιστική σφαιρική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις, τις προκλήσεις όπως είναι η κρίζωση της ε, φτώχειας, ε, ε, κακή διακυβέρνηση, οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία και μάλιστα όχι μόνο στο Μαλί αλλά σε όλο το Σαχέλ και τη γειτονική Λιβύη. Δεν πρόκειται να βοηθήσουμε μόνο το Μαλί αν δεν αναλάβουμε δέσμευση στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ. Για Ευχαριστώ, Πρόεδρε η επάνωδος του Μαλή στην κανονική πορεία μετά το πραξικόπημα παραμένει το ζητούμενο. Υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ε, η, η περιοχή του Κιντάλ δεν είναι ακόμη ασφαλής. Ε, και θα πρέπει και οι Τουαρέγκ να συμμετάσχουν στην εξέβρεση μιας λύσης. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ο ευάλωτο χαρακτήρας όλη τη περιοχή του Σαχέλ που εκτίθεται ε, σε ε, όλο τον αντίκτυπο της Αραβική άνοιξη. Όλα αυτά δεν θα πρέπει βέβαια να θεωρηθούν ότι έχουν ε, δώσει ένα τέλος στη βία στην περιοχή ο στρατός ετοιμάζεται να ε, ε, απειλήσει και πάλι ολόκληρη την περιοχή. Υπάρχει η ημερομηνία ε, του Ιουλίου ε, για τις ε, προεδρικές εκλογές και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει παρατηρητές στις εκλογές υπό την προεδρία του Λουί Μισελ που γνωρίζει την πραγματικότητα των... και την καθημερινότητα στις χώρες της Αφρικής και οι δυνάμεις ε, των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα παράδειγμα ε, όσον αφορά τις ειρηνευτικές ε, δυνάμεις. Είναι θετικά τα αποτελέσματα της σύσκεψης των δωρητών που έγιναν στις Βρυξέλλες το Μάιο που είναι έτοιμοι να δώσουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση της χώρας. Τώρα όσον αφορά το αν οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στην αρχή της ανασυγκρότησης του κράτους του Μάλι ή στο τέλος, εγώ είμαι πεπισμένος ότι η στο τελος εγω ειμαι πεπισμενο οτι η διεξαγωγη των προεδρικών εκλογών παρά τις αμφιβολίες που μπορούμε να έχουμε, όπως προανέφερα, είναι σωστή απόφαση και θα σας πω γιατί. Οι εκλογές εντάσσονται στη μακρά διαδικασία εκδημοκρατισμού του Μαλή που ήδη ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 το να οικοδομηθεί το κράτος πριν από τις εκλογές είναι κάτι το οποίο δεν θα λάμβανε υπόψη ότι μόνο η καθολική ψηφοφορία θα μπορούσε να νομιμοποιήσει ε, τα θεσμικά όργανα και να τους εξασφαλίσει την καλή λειτουργία θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη τους θεσμούς τους. Και κλείνοντας, θα ήθελα ε, να επιστήσω την προσοχή σας, κύριε Επίτροπε, στην άρνηση χορήγησης ε, θεώρηση διαβατηρίου στην κυρία Τραωρέ, πρώην Υπουργό Πολιτισμού στην Ευρώπη. Γνωρίζω την κυρία Τραωρέ εδώ και χρόνια και δεν θα μπορούσα να, σε καμία περίπτωση να φανταστώ ποιοι λόγοι οδήγησαν στο να της αρνηθούν τη θεώρηση διαβατηρίου. Για τους πράσινους Αλφόνση ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Μαλί είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε το Βόρειο Μαλί τους επόμενους ε, μήνες θα εξαρτηθεί για τα επόμενα 15 χρόνια η κατάσταση στην περιοχή αυτή. Υπάρχει ο κίνδυνος για μια σύραξη ε, ανάμεσα στους κατοίκους του Μαλή για λόγους εκδίκησης υπάρχει ένα πνεύμα πραξικοπηματικό και μετά από την γαλλική παρέμβαση δεν έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια αυτά. Όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη συνάντηση που θα έχουμε την επόμενη Δευτέρα θα το θέσουν το θέμα. Η στρατιωτική πρωτοβουλία, η επιτυχής εναντίον των τρομοκρατών και των εμπόρων ναρκωτικών δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο στρατιωτικής εισβολής του ε, Μαλή στο Κιντάλ και στο Αζαουάντα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ομοσπονδιακό κράτος με πραγματική αυτονομία που θα διασφαλίσει την ισορροπία και τη σταθερότητα της περιοχής αυτής για τους συντηρητικούς Τσαχράντιλ 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, διάβασα σήμερα μία έκθεση που δείχνει τι συνέβη στο Μαλί και τι καταστροφή έλαβε χώρα ε, στην Τιμποκτού για παράδειγμα Εκεί 16 σημαντικά μνημεία καταστράφηκαν, αναφέρει η UNESCO, και χιλιάδες χειρόγραφα κάηκαν. Πρόκειται για μια πολιτιστική καταστροφή τεραστίων διαστάσεων. Επίσης, σοβαρή όμως είναι η πολιτική και η οικονομική καταστροφή, που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, γιατί καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή. Είναι γνωστό ότι η ομάδα μου είναι πολύ επιφυλακτική απέναντι στις ευρωπαϊκές λύσεις. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ τάσομαι υπέρ της ανάμειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανέβρεση λύσης για το Μαλί. Και θα στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες και τις δράσεις που θα εξασφαλίσουν την κυριαρχία του Μαλί. Και επίσης ε, θα βοηθήσουν στην επανασυμφιλίωση. Αναφέρθηκε πολλές φορές ο ρόλος της ε, Γαλλίας και θα πρέπει να αναγνωριστεί γιατί κάποιος έπρεπε επιτέλους ε, να αναλάβει δράση σε διεθνές επίπεδο και αυτό το έκανε η Γαλλία. Επίσης ε, είναι σημαντική και η αποστολή κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τσεχία έχει στείλει 40 στρατιώτες στην περιοχή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να είμαστε δραστήριοι στην περιοχή αυτή. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ εκ μέρους της ΓΚΟΕ, η κυρία Λέζινγκ, για ένα λεπτό. Με τη στρατιωτική παρέμβαση προσπαθήσαμε να δώσουμε μια λύση. Δεν δόθηκε όμως καμία λύση. Απλώς ενισχύθηκε η αβεβαιότητα και η βία στην περιοχή. Πίσω από την κρίση βρίσκονται και διεθνείς παράγοντες που προκάλεσαν την έκρηξη της κρίσης και πίσω από αυτό βρίσκονται διάφορα συμφέροντα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της κρίσης και θα πρέπει να δούμε το διεθνές πλαίσιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και θα πρέπει τέλος να δούμε το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών στο οργανωμένο έγκλημα και στην πρόθεση ομάδων σαλαφιστών. Είναι μια πολιτική που δεν νομιμοποιείται διότι προσπαθεί να προωθήσει την εξόριξη ουρανίου ή και την δολοφονία παιδιών. Το Μαλί είναι μια πλούσια χώρα αλλά ο λαός παραμένει φτωχός και συνεχίζει να υποφέρει ενώ άλλοι πλουτίζουν εις βάρος τους. Η υπόλοιποι εγγεγραμμένοι στρίφλερ 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πήγα στο Μαλί εδώ και μια βδομάδα και στη Μαυριτανία επίσης η κατάσταση ανθρωπιστική στο βόρειο τμήμα της χώρας είναι ανησυχητική. Αποκρύβεται, σκιάζεται από τις εκλογές που είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και την διεθνή κοινότητα σε επίπεδο χρηματοδότησης. Η κατάσταση στα τρόφιμα χειροτερεύει. Η ενδιάμεση περίοδος η οποία ξεκινάει τώρα είναι πραγματικά επικίνδυνη και δυστυχώς θα οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων και σε επιδημίες όπως η χολέρα. Ο βοράς της χώρας παραμένει ένας χώρος ανεξέλεγκτος με ελεύθερους τσιχαντιστές και λαθρεμπόρους. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες λόγω της απουσίας των κρατικών δομών, αλλά όχι πάντα με επιτυχία. Πήγα στα στρατόπεδα Ανταρά στη Νότια Μαυριτανία και εξέφασα τις ανησυχίες μου για τις άσχημες συνθήκες και τις εντάσεις ε, στο στρατόπεδο αυτό. Ε, υπήρξε μια μεγάλη καταιγίδα πριν δύο εβδομάδες και δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα και θα συνεχιστεί αυτό γιατί οι πρόσφυγες δεν θέλουν να επιστρέψουν στο Μαλί όσο δεν διασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Οι εκλογές αυτές είναι βασικό βήμα βέβαια για την επιστροφή στη δημοκρατία. Η σωστή διεξαγωγή των εκλογών στο βόρειο κομμάτι της χώρας είναι βασικό πράγμα για την αξιοπιστία των εκλογών διαπίστωσα επιτόπου ότι υπάρχει πραγματική επιθυμία των αρχών των τοπικών για να γίνουν οι εκλογές. Παίζεται βέβαια και ιδιαίτερα λόγω των απειλών στον τομέα της ασφάλειας, της ψήφου των εκτοπισμένων και των προσφύγων και τα προβλήματα που έχει γενικά η διοίκηση στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Κιντάλ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι οι παρόντες ε, έχουμε επίγνωση της ε, δέσμευσης και της πολύ καλής προσπάθειας που κάνουμε στο Μαλί. Γνωρίζετε ότι είναι τεράστιες οι προκλήσεις, κοινέ και φυσικά θα πρέπει να μαγιστοποιήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και τη συνεργασία με το Μαλί. Αυτή τη στιγμή δίνουμε πολύ σημαντική βοήθεια σε μία από τις 10 φτωχότερες χώρες του κόσμου. Και σίγουρα 650.000 άνθρωποι χρειάζουν άμεση επιστηστική βοήθεια και 660.000 ε, παιδιά υποσυντίζονται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συντονισμό με τους υπόλοιπους δωρητές και κυρίως να συνεργαστούμε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται επί τόπου, ώστε να αποφύγουμε το λοιμό για χιλιάδες ανθρώπους. Συνεχίζονται δυστυχώς κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μένουν ατιμόρυτες, ε, ε, στρατολόγηση παιδιών, ε, βασανιστήρια, κρατήσει από άνθρωπες συνθήκες. Και ο άμαχος πληθυσμός ζει σε μια δύσκολη κατάσταση, κάτι που είναι ακόμη χειρότερο για γυναίκες και παιδιά. Πώς πρόκειται να ενισχύσετε το την βοήθειά μας και κυρίως να εξασφαλίσετε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μαλί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Ρινάλντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για το Μαλί. Έχουμε τρία θέματα. Το πρώτο είναι η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, δεύτερον είναι η στρογγύλη τράπεζα των δωρητριών χωρών και έχουμε επίσης και ένα θα έλεγα χρονολόγιο εκλογικό για τις προεδρικές και ίσως αργότερα τις βουλευτικές εκλογές. Ελπίζω να αντιμετωπίσουμε με ενωτικό τρόπο όλα αυτά τα θέματα μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στη Συρία. Το Μαλί παραμένει θύμα ενός πολέμου για το οποίο δεν ήταν υπεύθυνη η ίδια η χώρα. Υπήρχαν βάρβαροι που κατέστρεψαν τα πάντα, ε, έκοβαν χέρια, βίαζαν γυναίκες και κατέστρεφαν τα μνημεία του πολιτισμού όπως και στο Αφγανιστάν. Πρέπει να υπάρξει σωστός συντονισμός για να αποφύγουμε την κακοφωνία και τις επικαλύψεις από τους ε, ε, από τις δωρήτριες χώρες. Ε, οι χρηματοδοτήσεις τώρα ξεκίνησαν να έρχονται, να έρθουν πραγματικά. Και τρίτον θα πρέπει η πολιτική τάξη του Μαλή να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί το Μαλή είναι θύμα και των εσωτερικών του αντιφάσεων και αυτή η κρίση θα προσπαθήσει να ξεπεράσει κατά πολέμηση της διαφθοράς, κόμματα τα οποία να έχουν πραγματικούς εθνικούς στόχους και εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλο το έδαφος. Η ειρήνευση του βορρά της χώρας ε, έχει, είναι μια σωστή προσπάθεια. Ε, στο Μαλί λέγεται ότι καμιά ασθένεια δεν είναι φυσική, για, για τα πάντα φταίει κάποιος ή κάτι. Ε, είναι γνωστά τα ονόματα αυτών που προκάλεσαν προβλήματα στο κράτος δικαίου και στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτές, αυτά τα μαύρα μυαλά, όπως έλεγαν, θα πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε η πολιτική ε, τάξη του Μαλή να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Γκάλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανασυγκρότηση και ο δημοκρατισμός ε, στο Μαλί είναι κάτι το οποίο είναι προς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο του Μαλί. Δεν θέλουμε να υπάρξει ένα κενό στο Μαλή και στο Σαχέλ όπου να μπορεί να αναπτυχθούν ε, ε, εκπρόσωποι της Τζιχάντ ή άλλοι φονταμενταλιστές. Είναι σημαντικό λοιπόν και είναι σωστό ότι ε, παρενέβη η Γαλλία και ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποστείλει μια εκπαιδευτική αποστολή. Εκδημοκρατισμός σημαίνει και ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και πολλοί συνάδελφοι έθεσαν εδώ ένα ερωτηματικό. Και θα ήθελα να πω ότι και εγώ ως επικεφαλής της ομάδας παρατηρητών στην Τινησία και στο Πακιστάν γνωρίζω ε, τι πρέπει να κάνει κανείς να ξεκινάει από το μηδέν. Στην Τινησία ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και πρέπει να γίνουν οι εκλογές το Μάιο και τελικά κατάφεραν ούτε τον Ιούλιο αλλά τον Οκτώβριο να κάνουν τις εκλογές. Υπάρχουν όντω ερωτηματικά για το πόσο, κατά πόσο μπορούν να οργανωθούν εκλογές με τους κατοίκους του Μαλή που, ώστε να έχουμε μια θετική αξιολόγηση τελικά. Και ο συνάδελφος Λουί ε, Μισελ δεν μπορεί να εφεύρει κάποια διαφορετικά στάνταρτ και πρότυπα. Θα ακολουθήσει αυτά τα οποία γνωρίζουμε στην ευρωπαϊκή μας κοινότητα και τα διεθνή πρότυπα που ε, ισχύουν. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν εκλογικοί κατάλογοι που να αληθεύουν, όχι μόνο στο Τιμπουκτού, αλλά και σε όλες τις περιοχές του Μαλή και θα πρέπει οι εκλογείς να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να πληροφορηθούν για τους υποψηφίους. Θα πρέπει οι υποψήφοι να μπορούν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Όλες οι δομές θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορούμε στο τέλος να πούμε ναι όντως ήταν εκλογές που ανταποκρίνονται σε ένα επαρκές πρότυπο. Και εδώ βεβαίως και έχω κάποιες αμφιβολίες ε, και ελπίζω ότι μπορούμε μαζί με τις αρχές του Μαλή μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον να κάνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να μην υπάρχουν επιπλέον προβλήματα πέραν της ανασυγκρότησης, να μην ε, μπορούν να ισχυριστούν αυτοί οι οποίοι θα έχουν χάσει τις εκλογές ότι δεν ήταν δημοκρατικές οι εκλογές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τυρολιά για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η εδαφική ακαιρεότητα του Μαλή, η ανασυγκρότηση, η αναφορά της ειρήνης είναι σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ταχθεί στο πλευρό της Γαλλίας σε αυτή την κρίσιμη φάση. Η διεθνή σύσκεψη των δωρητών επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σχεδίου δράσης και εξασφάλισε με μεγάλες υποσχέσεις, 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι δυστυχώς που υστερεί σε σχέση με τις προσδοκίες μας, γιατί οι αρχές του Μαλή έχουν τεράστιες προκλήσεις. Είναι πολύ, πολύ έφραυστοι οι θεσμοί και υπάρχουν προβλήματα διακυβέρνησης. Κάτι που θα ε, πλήξει την αξιοπιστία του κράτους απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα στο Βορρά. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτή τη διαδικασία και οι εκλογές είναι πολύ σημαντικό γιατί οι μεταβατικές αρχές, η πρωτοβουλία των μεταβατικών αρχών να προσκαλέσουν ευρωπαϊκή αποστολή παρατήρηση εκλογών είναι πολύ θετικό βήμα. Επίσης σημαντική είναι ανάγκη να εμπλέξουμε στο έπακρο τους περιφερειακούς εταίρους στη διαδικασία σταθεροποίησης του Μαλή, γιατί η, η, η συμμετοχή του Σαχέλ είναι πολύ σημαντική στις εξελίξεις του Μαλή και θα πρέπει ε, η, σημαντική, η δική μας συμμετοχή να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες λύσεις και στο Μαλή και στο Σαχέλ, γιατί η ασφάλεια στην περιοχή θα επηρεάσει και τη δική μας ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τιάστινη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τους Γάλλους για την επιτυχή επιχείρησή τους ε, στο Μαλί για να διαλύσουν ε, το, την συμμαχία του Κατάφη, της Τζιχάτ και τρομοκρατικών δυνάμεων που έλαβαν ε, τον έλεγχο σημαντικών αστικών κέντρων το 2012. οι εξτρεμιστές δεν είχαν νικηθεί ακόμη και μόνο με στρατιωτικές λύσεις δεν πρόκειται να επιλύσουμε το πρόβλημα του Μαλή. Θέλουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη Μαλή. Θα πρέπει γι' αυτό να εκριζώσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και να δούμε ποιες είναι οι αιτίες αυτής της ριζοσπαστικοποίησης. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ρίζες της αστάθειας και της σύγκρουσης σε μια περίπλοκη χώρα όπως είναι το Μαλή. Οι ρίζες αυτές είναι πολύ βαθιές και εσωτερικές πηγές ανασφάλειας και κάποια θεσμική αδυναμία και διαφθορά έχουν συμβάλει στην κατάσταση αυτή. Η ενδημική φτώχεια και οι κοινωνικο οικονομικέ εντάσει επίση επιδεινώνουν την κατάσταση. Το θέμα σήμερα είναι πώ θα μειώσουμε την πολιτική διαφθορά και πώ θα διορθώσουμε τι αδυναμίες στι υποδομέ και στην παροχή δημοσίων αγαθών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καστέξ, η κυρία Καστέξ, συγγνώμη, για 1,5 λεπτό. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πριν από λίγους μήνες, πολλοί είχαμε πει ότι είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναλάβει μεγαλύτερη δέσμευση για να αποφύγει την κρίση στο Μαλή, ε, στο πλάι της Γαλλίας και της στρατιωτικής παρέμβασης. Τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε να επανέλθει η χώρα στη δημοκρατία και κυρίως να αποφύγουμε μια νέα κρίση. Όλοι οι λόγοι που οδήγησαν στην κρίση συνεχίζουν να υφίστανται. Αυτή η πρόληψη θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η Γαλλία θα αποβούν εις αν η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της πρόληψης της κρίσης δεν έχει ένα μαζικό χαρακτήρα δεν αρκούν αυτές οι προσπάθειες για τις εκλογές στις 28 Ιουλίου για τη σταθερότητα της χώρας. Θα πρέπει να δεσμευθούμε με πλήρη δέσμευση, όχι μόνο υπέρ της δημοκρατικής διαδικασίας, αλλά και για την πρόληψη μιας νέας κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Εγώ θα ήθελα να τις, να στην επιστροφή των εκτοπισμένων και προσφύγων και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, ιδιαίτερα στις ε, τρεις περιφέρειες του Βορρά. Είναι θέμα ασφάλειας, ασφάλειας με αλφα και εδαφικής ακαιρεότητας που είναι σημαντική για το Μαλί. Για τον εκδημοκρατισμό θα πρέπει πρώτα να διεκπαιρεώσουμε και την εκλογική διαδικασία και η νομιμοποίηση, η νομιμότητα και η αποδοχή του αποτελέσματος, του εκλογικού αποτελέσματος θα, ε, θα συνδυαστεί με μια ε, κρατική διαδικασία σε όλη την επικράτεια του μάλι. Επίσης θα πρέπει στις εκλογές να συμμετέχουν όλοι. Και το λέω αυτό γιατί το ισχύον εκλογικό σύστημα επιτρέπει τη συμμετοχή μόνο του 30% των δικαιο... όσων δικαιούνται να ψηφίσουν σε σχέση με τα δικά μας δεδομένα. Θα πρέπει να διορθωθεί λοιπόν αυτή η αδικία και να μπορούν όλοι να ψηφίζουν. Η παρουσία της ε, Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλή θα πρέπει να είναι μετρημένη και προσεκτική. Να γνωρίζουμε πού βαδίζουμε και να αποφύγουμε πατερναλιστικές ε, συμπεριφορές και αφιψηλού και ιδιαίτερα ε, βεβαιασμένες ε, αξιολογικές κρίσεις. Και φυσικά εκεί που θα πάμε να πάμε με ασφάλεια. Με ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Και όχι σε ένα τμήμα μόνο της χώρας αυτής. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Ζάλα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντισταθεί στο ριζοσπαστικό Ισλάμ και στην τρομοκρατία. Και το Μαλί είναι μια χώρα κλειδί για αυτή την προσπάθεια. Βασικό μας καθήκον θα πρέπει να είναι να μην αφήσουμε αυτό το φαινόμενο να εξαπλωθεί στην υποσαχάριο Αφρική. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να ισχύσει μια περιοχή ασφαλείας από ε, το Σαχέλ μέχρι το Σουδάν και στο κέρας της Αφρικής. Είναι αναπόφευκτο το ότι πρέπει να μας απασχολήσει ένας στρατηγικός μηχανισμός ασφάλειας που θα υλοποιηθεί σε αυτή την περιοχή και θα δημιουργήσει ένα φράγμα μεταξύ της υποσαχάριας Αφρικής και της Βορείου Αφρικής. Κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα μπορούμε να απαλλαγούμε από τα αρνητικά φαινόμενα και η σταθεροποίηση του Μαλή θα επιτευχθεί εάν μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό, κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως διαπιστώθηκε και στη διάσκεψη για το Μαλή το Φεβρουάριο φέτος ε, υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αφήσει τους κατοίκους του Μαλή να πρωταγωνιστήσουν στην ανέβρεση ειρηνικής λύσης από την κρίση και να μπορέσουν όλοι να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να αποφύγουμε μεμονωμένες πολιτικές για την εξάρθρωση της τρομοκρατίας και της ρεσουστικοποίησης, γιατί ο λοιμός η ξηρασία και η αδυναμία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει επιστηστική ασφάλεια δημιουργεί δυσαρέσκεια και απογοήτευση στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει οικονομική και πολιτική βοηθεία στην ε, πρωτοβουλία του Σαχέλ ως τμήμα μια συνολικής προσπάθειας να, να καταπολεμηθούν τα αίτια των προβλημάτων του Μαλή για να βοηθήσουμε το Μαλί να επαναφέρει τη σταθερότητα και να αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη ζητήματα της επιστικής ασφάλειας σε συνδυασμό με την κατάρτιση του στρατού του Μαλί θα έχουμε τα πρώτα βήματα στο σωστό δρόμο. Χαίρομαι για την εγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αποστολής για την κατάρτιση των στρατευμάτων του μαλί κάτι που θα συμβάλλει στην ε, μεγαλύτερη ασφάλεια της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και να βοηθήσει τους κατοίκους του Μαλή να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ευχαριστώ. E Ο κύριος Γκάμπριελ, 1,5 λεπτό. Η κυρία Γκάμπριελ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση στο Μαλί παραμένει ε, πολύπλοκη και οι συζητήσει στο Μπουκάμπε μαζί με ε, τον πρόεδρο Μπουρκίνα Μπέ είναι αποφασιστικέ. Οι εκλογέ προβλέπονται για τι 28 Ιουλίου και μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση του Μαλί. Είναι πολύ σημαντικό να μην γίνουν αντιπαραγωγικέ αυτέ οι εκλογέ. Θα πρέπει να είναι ασφαλεί και αυτό είναι βασικό ζήτημα. Ε, αυτό είναι απαραίτητο και για την αποστολή εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, και να πρέπει να έχουμε κατά νου τα διδάγματα του Μαρτίου του 2012. Μία συμφωνία για την ε, επάνωδο στην ειρήνη των ε, δυνάμεων του Μαλή είναι επίση ένα θετικό σήμα γιατί πρέπει ο στρατός να εγγυάται την ακαιρεότητα του, της επικράτειας ε, του Μαλλιού όπου θα γίνουν οι εκλογές. Και όπως είπατε κύριε Επίτροπε, η διεθνής κοινότητα, ο Γαλλικός στρατός και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μίνουσμα δεν μπορούν παρά να είναι συνοδευτικά για αυτή την ασφάλεια της επικράτειας. Δεν μπορούμε εμείς να υποκαταστήσουμε το κράτος του μαλί. Επίσης, για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, όλα τα σημερινά προβλήματα δεν μπορούμε να τα αναβάλουμε για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ανάμεσα στα υπόλοιπα κατεπήγοντα θα πρέπει κάθε μορφή βίας κατά του πληθυσμού, του άμαχου πληθυσμού ε, να ε, την χάνουν συνέχεια. Χρειάζεται αποστολή παρατήρηση των εκλογών, χρειάζεται επιρογνωμοσύνη για το χάρτη πορεία για το Μαλί και όλα αυτά θα αποδείξουν τη δέσμευσή μα υπέρ του Μαλί. Η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετεκλογική περίοδο που τη έχουμε υποσχεθεί θα είναι αποφασιστικό και θα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μα. Για την ανάπτυξη στο Σαχέλ θα πρέπει να ενισχύσουμε όλη αυτή την περιοχή για να συνεισφέρουμε στην σταθεροποίηση όλης της περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ. Η κυρία Κόρχολα. Εδώ και ένα χρόνο αναφέρθηκα στην κατάσταση στο Μαλί, στην αίθουσα αυτή και ζήτησα να υπάρξει διάλογος έτσι ώστε να γίνουν διαπραγματεύσεις στις αρχές του 2013 δημιουργήθηκε μια επιτροπή συμφιλίωσης, μια επιτροπή διαλόγου, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν μόνο φυσικά μια συνεννόηση σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά απαιτούν και βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει την χώρα αυτή και θα πρέπει η προσπάθεια αυτή οικονομική να ενισχυθεί και να βοηθήσουμε στην διασφάλιση της χώρας. Θα πρέπει όλες οι ένοπλες πλευρές να συμμετέχουν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης έτσι ώστε οι ελπίδες και οι ανησυχίες τους να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίμπαλξ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, έγινε μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση και γι' αυτό θα επαναλάβω κάποια σημεία που μου φαίνονται κρίσιμα. Καταρχάς, η υποστήριξη προς το Μαλί γίνεται υπό την αιγίδα της ίδιας της χώρας. Εμείς υποστηρίζουμε τον οδικό χάρτη που ε, διατυπώθηκε από τις αρχές του Μαλί και επίσης ε, ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μέχρι το 2014 που διατύπωσαν οι ίδιοι. Το Μαλί είναι υπεύθυνο για τις εκλογές, υποστηρίζουμε την προσπάθεια μέσω της αυμόδιας υπηρεσίας ε, των Ηνωμένων Εθνών και ελπίζουμε οι εκλογές αυτές να είναι αξιόπιστες και δημοκρατικές και όλοι να πάρουν μέρος σε αυτές. Δεύτερον, Ίσως ε, δεν αναφερθήκαμε επίσης στις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μια δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναπτυχθεί Νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη θα είναι καθοριστική. Το τρίτο θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι ε, μορφής αλληλεγγύη υπάρχει προς τους κατοίκους του Μαλή. Η υπόσχεση προς υποστήριξη βέβαια δεν προέρχεται μόνο από τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από ε, μια ε, ομάδα εκπαίδευσης η οποία προέρχεται από τη Λετωνία και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και υποστηρίζεται από το λαό της Λετωνίας. Έχουμε υπογράψει και μια οικονομική συμφωνία με το Μαλί για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας των πολιτών. Και τέλος, σε τεχνικό επίπεδο μαθαίνουμε πώς να εργαζόμαστε σωστά στο ΣΑΕΛ. Το ΣΑΕΛ είναι μια δύσκολη περιοχή και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία στο ΣΑΕΛ που διαμορφώθηκε το 2011 είναι μια καλή βάση και η έκθεση ελέγχου προτείνει κάποια επιπλέον στοιχεία. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια καλή βάση και δίνει δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί Έχουμε περιορισμένα οικονομικά μέσα και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο και να υποστηρίζουμε δραστηριότητες που θα καταστήσουν το ΣΑΕΛ πιο σταθερό και πιο ευήμερο μακροπρόθεσμα. Τέλος, μια προσωπική παρατήρηση. Αποτύχαμε ή όχι στην αναπτυξιακή συνεργασία με το Μαλί. Θυμάμαι τον πρόεδρό μου να μιλάει σε αυτό εδώ το σώμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια εύθραστη χώρα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε να την υποστηρίξουμε στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της ανάπτυξης. Δεν είχαμε προβλέψει τη στρατιωτική σύγκρουση, αλλά ακόμα και αν το είχαμε προβλέψει, τι θα μπορούσαμε να κάναμε. Γιατί ακριβώς ε, η αποστολή εκπαίδευσης που έχουμε στείλει ε, γίνεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης. Ε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη, υπάρχουν όρια σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε, σε σχέση με το βορρά, σε σχέση με τις απειλές, αλλά είναι μια χώρα με μια νόμιμη κυβέρνηση και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς τις απόψεις μας. Είναι λοιπόν δύσκολο να συζητιούνται κάποια θέματα με τέτοιο τρόπο και κάποια θέματα τα οποία η κυβέρνηση δεν θα έλεγα φροντίζει να τα καλύπτουμε εμείς. Υπήρξαν όρια λοιπόν στη συνεργασία με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του Μαλή, μας έθεταν ορισμένα όρια, αν ήμασταν πιο θαραλέοι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τη στρατιωτική κρίση. Αλλά αυτά γνωρίζαμε, αυτά κάναμε στη δεδομένη στιγμή. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το τι κάναμε, για το τι κάνουμε και μπορούμε τεχνικά να βελτιώσουμε την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ Επίτροπε. Έχω λάβει λοιπόν την πρόταση ψηφίσματος που κλείνει την συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι.